πρακτικά. Πριν περάσουμε στην συζήτηση έχω τρεις ανακοινώσεις να κάνω. Η πρώτη, όπως ε, θα θυμάστε, ο πρόεδρος της 9 2016 έλαβε άμεσα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 165 παράγραφος 3 ε, σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του κανονισμού και απέβαλε τον κύριο Συναδεινό από το υπόλοιπο της συνεδρίασης για τις απαράδεκτες παρατηρήσεις του για τον τουρκικό πληθυσμό. Μετά από ακρόαση του κυρίου Συναδεινού και σύμφωνα με το άρθρο 166 του κανονισμού, ο πρόεδρος αποφάσισε να επιβάλει κύρωση κατά του κυρίου Συναδεινού, η οποία είναι στέρηση της μερίσχες αποζημίωσης για μια περίοδο 10 ημερών και κοινοποιήθηκε η απόφαση σήμερα στον ε, κύριο Συναδεινό. Δεύτερη ανακοίνωση. Η κυρία Τζέιν Κόλινς ζήτησε